δεν θα γίνει αύριο. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι μια προφορική ερώτηση για την απαιτούμενη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την πρόσβαση στα έγγραφα μετά τη θέση ενισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Μάικλ Κάσμα που είναι ο εισηγητή. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι χαίρομαι που βλέπω την Επιτροπή Βόλστρομ στην ε, Θούσα και την Σεσίλια Μάλστρομ που είναι η Προεδρεύουσα γιατί από το 99 ήδη από την αρχή του εξέδωση του κειμένου αυτό έχουμε ασχοληθεί με το θέμα. Είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτό που πετύχαμε τον Μάη του 2001 ήταν μια ιστορική ε, επιτυχία μεταξύ πολλών χωρών, 15 χωρών που ερχόντουσαν από διαφορετική, διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικές συνήθειες να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για τη διαφάνεια και αυτό σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην αποφασιστικότητα της τότε Σουηδικής Προεδρίας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οφείλεται επίση την αποφασιστικότητα τη Εκτελεστική Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι και τα τρία θεσμικά όργανα χρειάζονται ε, μια πολιτιστική αλλαγή έπρεπε να πούμε ότι το άνοιγμα και η διαφάνεια δεν θα πρέπει να αποτρέψουν ε, την ε, δημοκρατία των εντύων. Τις επιτρέπουν να θύσει γιατί επιτρέπει στους πολίτες να δουν τι γίνεται στο όνομά τους. Και αυτό μας επιτρέπει να σηκώσουμε το πέπλο για να δει ο καθένας ότι δεν υπάρχουν τεράστια μυστικά ούτε στο Συμβούλιο ούτε στην Κομισιόν. Για το Κοινοβούλιο δεν είμαι πολύ σίγουρος αλλά ελπίζω ότι και στο Κοινοβούλιο έχει στα υπόγεια του κάποια μυστικά. Θα ήθελα λοιπόν ευχαριστήσω την Επίτροπο και να αναφερθώ και στην αγαπητή συνάδελφο Σασίλια Μάλστρομ που κατέβαλε τις προσπάθειες αυτές. Τώρα χρειαζόμαστε μια άλλη δέσμευση. Όπως είπα, πολλά πετύχαμε, πάρα πολλά. Έχουμε ένα κατάλογο των εγγράφων, έχουμε στην ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ορίζουμε και επανορίζουμε αυτό που είχε συμφωνηθεί αρχικά για την πρόσβαση στα έγγραφα. Αποδεχόμαστε ότι όλα τα έγγραφα θα πρέπει να παραμείνουν προσβατά. Και αν δεν είναι προσβατά θα πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση γιατί δεν είναι προσβατά. όσον αφορά το άρθρο 4 για τις εξαιρέσεις ή το άρθρο 9 για τα ε, απορρίτα έγγραφα. Τώρα όμως η Κορεπέρ έχει και ζητήσει μια αναθεώρηση. Ξέρω ότι εδώ έχουμε διαφορετικές απόψεις γιατί η αναθεώρηση έγινε με υποβολή στο Κοινοβούλιο. Είχαμε την πρώτη ανάγνωση το Μάρτιο φέτος και αυτή η μεταρρύθμιση που προέβλεπε η Κομισιόν δεν πήγαινε αρκετά μακριά. Έχουμε την εντύπωση ότι υπήρχε μια προσπάθεια να μειωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα. Ιδίως στον επανορισμό των εγγράφων, η ιδέα ότι θα πρέπει να εξαιρούνται κάποια, ε, κάποια έγγραφα και η έννοια του βέτο του, των τρίτων οι επισκέπτες που είναι εδώ απάνω στα θεωρία θα νομίζουν ότι κάτι που συζητάμε ήταν κάτι που έγινε στο διάστημα. Αυτό που συζητάμε όμως είναι ένας νόμος που τους επιτρέπει να ελέγχουν ότι είμαστε υπόλογοι. Εμείς, ως βουλευτές, είμαστε υπόλογοι για αυτά που κάνουμε στο όνομά τους. Και η Κομισιόν το ίδιο. Και το ίδιο και το Συμβούλιο. Πώς να γίνεται αυτό και το κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις εάν το τι κάνει ποιος παραμένει απόρριτο. Και ανοίγει μονάχα εκείνους τους εκπροσώπους λόμπι και δικηγόρους που ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Αυτό λέει ακριβώς η συνθήκη της Λισαβόνας. Λέει ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουν τη δημοκρατία, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στα έγγραφα, και γι' αυτό καλούμεθα να υπάρχει μια σειρά νέων μέτρων για την πρόσβαση. Βασικό όμω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα που υπάρχουν ήδη δεν θα μειωθούν και να γνωρίσουμε ότι μέσα στα πλαίσια τη Λισαβόνη δεν είναι μόνο τα τρία θεσμικά όργανα αλλά όλε οι υπηρεσίε, όλα τα σώματα που έχουν οριστεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παραδείγματο χάρη, καμιά φορά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπόλ, η Eurojust όλα αυτά τα όργανα είναι τώρα πια υπόλογα μέσα στα πλαίσια του κανονισμού 1049. Και πιστεύουμε οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τότε που τέθησε ισχύ η συνθήκη της αγώνας δεν είναι σύμφωνες ούτε με το πνεύμα ούτε με το γράμμα της συνθήκης αυτής ή με τις υποχρεώσεις που πιστεύουμε ότι συμπεριλαμβάνονται μέσα στα πλαίσια του κανονισμού 1049 2001 που προβλέπει απρόσβατη του κοινού σε όλα τα έγγραφα που προετοιμάζουν τα τρία θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. I thank you, Mr. Cashman. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κάσμαν και κύριε Μάλσον για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μέσω του Μάικλ Κάσμαν έθεσε αυτή την προφορική ερώτηση. Όπως ξέρετε, η διαφάνεια είναι θέμα ιδιαίτερα προσφυλές και στην Σουηδική Προεδρία. Και διανύσαμε μεγάλο δρόμο τα θεσμικά όργανα στον τομέα της διαφάνειας. Η διαφάνεια όμως δεν είναι μόνο θέμα διατάξεων, αλλά θέμα και νοοτροπίας και συμπεριφοράς και έμπρακτης εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων. Σήμερα το πρωί είχα τη χαρά να συναντήσω την Μάργαρετ Βάλστρομ και την Diana Wallis στην Διοργανική Επιτροπή για την πρόσβαση στα έγγραφα. Πρόκειται για μια επιτροπή που είχε να συνεδριάσει εδώ και δύο χρόνια. Είχαμε πολύ συγκεκριμένες συζητήσεις ε, προκειμένου να βελτιώσουμε την ε, πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινοτικά όργανα και θα πρέπει να συνεδριάζουμε πιο συχνά. Αυτό ήταν το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε. Η συνθήκη τη Λισαβόνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα τη διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι το καλύτερο μέσο για την πραγμάτωση τη δημοκρατία. Και μάλιστα ο κανονισμό 1049 αυτό το θέμα διέπει την πρόσβαση στα έγγραφα και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και το άρθρο 15 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας που επιμένει στο θέμα της διαφάνειας και της ε, πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα. Στο παρελθόν, μόνο το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσαν ε, να, να ανοίξουν τα έγγραφά τους και προς πολίτες. Σήμερα το ευρύ κοινό έχει ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση σε όλα τα κοινοτικά έγγραφα αυτά που προέρχονται από τα θεσμικά και τα άλλα όργανα. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τα έγγραφα του Ελεκτικού Συνεδρίου, του ΔΕΚ και της Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά γενικώ ε, έχει διευρυνθεί κατά πολύ η πρόσβαση στα έγγραφα από τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στις νέες διατάξεις της συνθήκης και το Συμβούλιο με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο του 2008, το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις εργασίες του. Και μάλιστα έκτοτε μια ειδική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου συνεδρίασε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους για να καταλήξει σε κάποιες τεχνικές διατάξεις με βάση τις τροπολογίες που έχει υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Μάιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει να μην ε, καταλήξει συμπεράσματα και μάλιστα η Υπουργός Δικαιοσύνης ε, της Σουηδίας, η κυρία Άσκ, εμφανίστηκε στις 2 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και δήλωσε προθυμία για περαιτέρω συζήτηση στα θέματα αυτά και επίσης ε, εξέφρασε την προθυμία της να εξετάσει όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εμβαθύνουμε στο θέμα της διαφάνειας. Μέχρι στιγμής όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε την ευκαιρία να εξετάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερο ε, αναφέρθηκε στην επίπτωση της συνθήκη της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσει και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συνεχίσουμε τις ε, διαθεσμικές συζητήσεις προκειμένου να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο η νέα συνθήκη. Το άρθρο 15, παράγραφος 3 της συνθήκης αποτελεί την, την κατάλληλη νομική βάση που διέπει την πρόσβαση στα έγγραφα. Τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν την ενημέρωση των πολιτών, την σωστή πληροφόρηση. Πρόκειται για σημαντικά άρθρα για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και για την ενίσχυση της νομιμοποίησής τους. Μπορούμε να συζητήσουμε για τον τρόπο υλοποίηση των στόχων μας, αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι όλα αυτά τα άρθρα σχετίζονται με τη διαφάνεια. Νομίζω ότι περισσότερο θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα της πρόσβασης των εγγράφων από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ, η κυρία Βάλστρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Κύριε Κάσμαν, πρώτα απ' όλα απευθύνομαι σε εσά. Νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία δυνατότητα που μου προσφέρετε. Εγώ να ευχαριστήσω εσάς, γιατί εσείς ε, πραγματικά είσαστε, προσωποποιείτε τον αγώνα για αυτό τον κανονισμό για να ανοίξει το Κοινοβούλιο για να υπάρχει διαφάνεια. Είσαστε, αν θέλετε, το σύμβολο, ο υπέρμαχος όλης αυτής ε, της, της, ε, της μάχης. Επίσης ε, και η κυρία Μάλστρομ και εγώ έχουμε αγωνιστεί για αυτή την υπόθεση και κανείς δεν αμφισβητεί ότι θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Ε, βέβαια, ε, παίζουμε διαφορετικούς ρόλους ε, και αναγκαστικά ήρθαμε σε σύγκρουση. Μερικές φορές ε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο τι μπορούμε να επιτύχουμε. Υπήρξε λοιπόν μια διαμάχη ανάμεσα στους ε, θεσμούς και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Ε, το πολιτικό κλίμα έχει αλλάξει, η πολιτική ισορροπία έχει αλλάξει και αυτή και τούτο λοιπόν έχει αναπόφευκτα επηρεάζει και τις συζητήσεις μας επί του θέματος. Όμως θα έλεγα ότι το σημείο κίνησης είναι ακριβώς το ίδιο. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι ειδικά αυτός ο κανισμός για την πρόσβαση στα έγγραφα μας εξυπηρέτησε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών αποδείχθηκε ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και άλλοι, πολύ περισσότεροι από αυτούς ε, που πληρώνουν για να το πράττουν από τους εκπροσώπους ομάδων πιέσεων που θέλουν να έχουν τα έγγραφα στα χέρια τους. Εμείς θέλουμε το κοινό, οι δημοσιογράφοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τα έγγραφα, να έχουν απόλυτη πρόσβαση σε αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο κίνησης για μένα ε, και γνωρίζω πολύ καλά ότι την άποψη αυτή και η κυρία Υπουργό. Βεβαίω η Σουηδική Προεδρία ήταν μια χρυσή ευκαιρία για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Τώρα λοιπόν θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που προσέφερε να λάβει χώρα αυτή η συζήτηση για τη διαφάνεια και για την καινούργια συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα δίνεται μεγαλύτερη σημασία σε αυτό που είναι ανοιχτό, που μπορεί να είναι ανοιχτό στη συμμετοχική ε, δημοκρατία. Και αυτή είναι η πλέον ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Τι είδους μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον κανονισμό 1049 του 2001. Και εξ όσων γνωρίζετε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας, εκεί που γίνεται λόγος για την πρόσβαση στα έγγραφα, τώρα πλέον η πρόσβαση επεκτείνεται και στα έγγραφα όλων των ε, οργάνων και των τομέων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για την Κεντρική Τράπεζα και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εθνικού λόγου. Όσον αφορά την αναθεώρηση του 1049 θα ήθελα να επισημάνω ότι η νέα νομική βάση το άρθρο 15 παράγραφο 3 τη συνθήκη που αφορά στη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το άρθρο μοιάζει με το παλαιότερο το το 2,55 και η κύρια διαφορά είναι ότι διευρύνεται ε, το πεδίο εφαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 ε, Δεκεμβρίου του 2009 προέβησε ανακοίνωση με στόχο του να προσαρμοστούν οι προτάσεις για δευτερογενή νομοθεσία σε σχέση με τη νέα συνθήκη. Όσοι βρίσκεστε εδώ γνωρίζετε την ε, ειδική γλώσσα που χρησιμοποιούμε και θα ξέρετε τον περίφημο νόμο λεωφορείο Omnibus Act. Ξέρετε ότι έχουμε εντάξει και ένα, μια νέα διάταξη έτσι ώστε να απευθύνει τη διαφάνεια και στους άλλους ε, στα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα. Αυτή η διάταξη έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η περαιτέρω πρόοδο στην νομοθετική διαδικασία οδήγησε στην έγκριση θα οδηγήσει μάλλον στην έγκριση του κανονισμού που βρίσκεται πλέον στα χέρια ε, του Κοινοβουλίου. Είμαστε στην πρώτη ανάγνωση. Ακόμα δεν έχουμε ε, καταλήξει νομοθετικά και δεν έχουμε και τη θέση του ε, νέου κοινοβουλίου. Βεβαίω και η Επιτροπή θα προχωρήσει, θα συνεχίσει για να επιτευχθεί συμφωνία ε, καθότι έχει ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία. Η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ένα ε, νομοθετικό πλαίσιο για τη συμμετοχική διαδικασία. Εμείς από πλευράς Κομισιόν ήδη έχουμε λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση των διαβουλεύσεων και τη συμμετοχή σε ε, συγκεκριμένες πολιτικές. Θα αξιολογήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές Κομισιόν για διαπραγματεύσεις με βάση τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας και θα αποφασίσουμε κατά πόσο είναι απαραίτητο να υπάρξουν προσαρμογές για βελτίωση. Και ξεκινήσαμε και να ασχολούμεθα με τις πρωτοβουλίε των πολιτών. Ακούμε τους πολίτες και τους άμεσα ενδιαφερόμενους πριν ε, καταθέσουμε πρόταση. Η μεγάλη σημασία που έχει η πρωτοβουλία των πολιτών αναγνωρίστηκε επίσης και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Η επερχόμενη Ισπανική Προεδρία, εξ όσων γνωρίζω, το θέμα αυτό το έχει βάλει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές της και θέλει να διεκπαιρωθεί ταχύτατα. Σήμερα το πρωί ακούσαμε τη Διοργανική Επιτροπή για την πρόσβαση στα έγγραφα αυτή συνήλθε μετά από πρόσκληση της Σουηδικής Προεδρίας έχει ως καθήκον να εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές το, να εξετάσει το ενδεχόμενο των ε, συγκρούσεων και την πρόσβαση στα έγγραφα. Αποφασίσαμε ότι θα έχουμε ε, μια ανοιχτή πύλη θα ε, έχουμε συμπληρωματικότητα των καταλόγων και επίσης θα προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τις προσπάθειες πρόσβασης. Εξάλλου θα ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις της πρόσβασης στα έγγραφα οποτεδήποτε δημιουργούνται ηλεκτρονικά αρχεία. Γνωρίζω ότι τέτοια εποχή του χρόνου ε, γράφεται και γράφουμε όλοι μας ε, τον ε, κατάλογο με τις ευχές μας. Όταν μιλάμε για την διαφάνεια και για το άνοιγμα, δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε στον Άγιο Βασίλη. Εμείς πλέον είμαστε αρμόδιοι να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις, να είμαστε σαφείς. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Προσβλέπω μεγάλη χαρά στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βέρστρα. Έχουμε τους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτη στο η κυρία Ζόμερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είχαμε συνεργαθεί με τους σκιώδεις των άλλων ομάδων και με τον εισηγητή να έχουμε μια προφορική ερώτηση. Ξεκινώντας από την απάντηση του Συμβουλίου και της Κομισιόν θα αποφασίσαμε το τι θα κάνουμε παρατέρω. Αυτή την απάντηση μάλλον μόλις την πήραμε γιατί ο εισηγητές εν αντιθέσει προς τη συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων ξαφνικά υπέβαλε ένα ψήφισμα το οποίο προτρέχει της δικής του άποψης και του του θέλει να έχει δηλαδή σαν απάντηση από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε και αυτό κύριε Κούσμαν έγινε μυστικά απόρριτο και χωρίς καθόλου διαφάνεια. Εσείς είπατε ότι είστε υπέρ της διαφάνειας, εσείς προσπαθήσατε να μας αφήσετε μας κατά μέρο. Και εκτός αυτού θα πρέπει να δούμε όσον αφορά το αποδεκτό αυτού του ψηφίσματος βάσει του καταστατικού. Γιατί επαναλαμβάνεται μια έκθεση που υπήρχε στο παρελθόν και είναι γι' αυτό περιττή. Ξέρω ότι είχαμε προσπαθήσει να πετύχουμε να υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα με του σκιώδες. Εγώ όμω είμαι κατά του ψηφίσματος. Με τη θέση ισχύει τη συνθήκη του Λισαβόνα κατά τη γνώμη μου, δεν τροποποιήθηκε τόσο πολύ η νομική βάση του θέματος που να προτροποποιεί τη δική μας θέση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί η έκθεση ήταν και είναι ένα θέμα που βασίζεται στην συναπόφαση και γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι η ομάδα μου αμφισβητεί το κατά πόσο είναι αποδεκτό σύμφωνα με τον κανονισμό το ψήφισμα. Δεν θέλω τώρα να περιπλάξω, περιπλέξω πάρα πολλά θέματα. Εδώ έχουμε αναφορές στο, στη συνθήκη της Λισαβόνης, στον χάρτα βασικών δικαιωμάτων και ούτω καθεστής για να νομιμοποιήσετε κάπως την πρόταση ψηφίσματος που υποβάλλετε. Αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό νομικά δεν είναι αποδεκτό. Λείπει μία αποδοχή ενός συμβαστικού χαρακτήρα που είναι μία εκ των ουσάνευ προϋπόθεση μέσα στα πλαίσια συμφωνιών με άλλες χώρες, παραδείγματο χάρη τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για το ΣΥΦΤΕ. Δεν υπάρχει και μία μεταβατική ε, λύση. Προσοχή των χρόνων, λέει ο Πρόεδρος. Και το θέμα τη ε, προστασία τη ιδιωτική ζωή, επίση παραβλέπεται. Θα πρέπει νομίζω αυτό το ψήφισμα να μην το ψηφίσουμε. Πήραμε μια καλή απάντηση από το Συμβουλίο και την Κομισιόν και θα μπορούμε βάσει αυτό να συνεχίσουμε την εργασία μα. Αυτό ήταν και ο στόχο τη προφορική μα. ερώτηση. Παρακαλώ, αποσύρατε την πρόταση ψηφίσματος τη, κυρία Κούσνα. Για δύο λεπτά η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, συμφωνώ με τον κύριο Κάσμαν που μας λέει ότι τώρα που έχει τεθεί σε ισχύ η συνδίκη της Λισαβόνης και υπάρχει μια νέα νομική βάση, είναι σωστό να έχουμε μια νέα συζήτηση του κανονισμού 1049 του 2001 όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συμβουλίου της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Η στήριξη της αγώνας έχει σαν στόχο να είναι πιο ανοιχτή η πρόσβαση και έτσι να είμαστε πιο κατανοητοί προς τους πολίτες. Γιατί η κατανόηση των πολιτών για την εργασία μας προκαθορίζει την, ε, το κατά πόσο πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η δυνατότητα οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, γι' αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική και ο κανόνας και το απαραίτητο να είναι μόνο η εξαίρεση. Τον Μάρτιο φέτος προετοιμάστηκε μια έκθεση για την πρόταση της Κομισιόν να τροποποιηθεί ο κανονισμός και αυτή η συγκεκριμένη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποτελέσει μια βάση για περαιτέρω συζητήσει. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συστάμε και στροπολογίε για τον οργανισμό που προποθέτει περισσότερο συνεργασία και κοινή συνένεση και των τριών θεσμικών οργάνων για την μεταρρύθμιση του ρόλου του στα πλαίσια τη διαφάνεια. Οι βελτιώσει. Αυτές θα δώσουν ε, ένα πολύ υψηλό επίπεδο διαφάνειας και θα επιτρέψει στους πολίτες να παρακολουθούν τις δημοκρατικές συζητήσεις και έτσι θα μπορέσουμε να ε, ε, κατανοηθούν συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό ζητώ από την Κομισιόν να τροποποιήσει τον κανονισμό των γλυκορότερο δυνατών και να επιτύχει μια κοινή θέση με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε εμείς να εξασφαλίσουμε ανοιχτό και συνεπή διάλογο με τους πολίτες. Η κυρία Νταϊάννα Γουόλης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ερώτηση και είμαι ευγνώμων προς τον κύριο Κάσμαν που μας παρουσίασε τις απόψεις του. Και είχα την εντύπωση ότι όλες οι πολιτικές ομάδες είχαν συμφωνήσει για το ψήφισμα. Αυτό εγώ είχα καταλάβει ως έκβαση της τελευταίας απογευματινής συνεννόησης των πολιτικών ομάδων. Μετά τη θέση ισχύ της ηθίκης της Λισαβόνας, χρειαζόμαστε μια ποιοτική αλλαγή στο όλο θέμα της διαφάνειας. Και ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδια για θέματα διαφάνειας, δεν τα έβρισκα πάντα εύκολα, αλλά Πιστεύω ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα έγγραφα και στην ενημέρωση. Είχα συνάντηση το πρωί με τη Σεσίλια Μάλστρομ και την κυρία Βάλστρομ που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Οπότε για πρώτη φορά τα τρία θεσμικά όργανα μπόρεσαν και συζήτησαν το θέμα και σημείωσαν πρόοδο. Αναφέρθηκε αυτή η σημαντική επιτυχία και καμπή. Δεν ε, δυνατό να συναντιόμαστε κάθε δύο-τρία χρόνια. Θέσαμε ήδη ημερομηνία για την επόμενη μας συνάντηση μέσα σε ένα εξάμεινο και με πιο τακτικό και συχνό χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα της δέσμευσής μας υπέρ της διαφάνειας και του ποιοτικού άλματος που πραγματοποιήσαμε σε αυτό το θέμα. Γιατί θέλουμε οι πολίτες μας να αντιληφθούν ε, όλα τα στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και να μπορούν να έχουν ε, ε, λόγο αλλά και εποπτεία της όλης αυτής της διαδικασίας. Νομίζω ότι και η δική ομάδα αλλά και όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν για κάποιες τροπολογίες που αντικατοπτρίζουν αυτή την πρόοδο. Ε, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ γιατί χάρη σε εμά τις τρεις κυρίες επιτεύχθη πρόοδο στο σημαντικό αυτό θέμα. Τρεις λοιπόν κυρίες και ένας κύριος που κάθεται εκεί, επάνω, επόμενος ομιλητής. Για ένα λεπτό κύριε Ζόμπρο. Κατά τη γνώμη πολλών ειδικών για τα νομικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά χρόνια στα θεσμικά όργανα αναφέρθηκε ίσως αβάσιμα η μορφή του δημοκρατικού ελλείμματος αναφέρθηκε τότε ότι πολύ σημαντικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται από ανώνυμους υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνονται κάπου μακριά στις Βρυξέλλες και μάλιστα με αδιαφανή τρόπο. Φάνηκε λοιπόν ότι η διαφάνεια είναι σημαντικό στοιχείο και θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι υπόλογα και υπεύθυνα απέναντι στην κοινωνία. Γιατί η ιστορία μας έχει διδάξει ότι αν δεν είναι υπόλογοι απέναντι στο κοινό, η εξουσία απαξιώνεται. Είχαμε παρόμοιε εμπειρίε στι διάφορε χώρε. Γι' αυτό και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι υπόλογα απέναντι στου πολίτε όλων των χωρών μελών. Και θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχή έλεγχο των αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα εξασφαλιστεί με την πρόσβαση στα έγγραφα. Στα έγγραφα εργασία, στι αναλύσει, στι μελέτε που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο. Επίσης, οι ομάδες πίεσης θα πρέπει, όταν ασχολούνται με ένα θέμα θα πρέπει να είναι διαφανής ο τρόπος της δραστηριότητας τους. Μόνο να είστε εξασφαλιστεί δημοκρατικός έλεγχος για όλους τους πολίτες όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και όλες τις οργανώσεις πολιτών, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους δημοσιογράφους. Έτσι, έχει εξαντληθεί ο χρόνος σας κύριε Σόμπρο θα πρέπει οι πολίτες να πιστούν ότι και οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά της όργανα ενδιαφέρονται για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Σταβάρης, για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, στο επίκεντρο τη συζήτηση βρίσκεται το θέμα τη εμπιστοσύνη. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κάθε στιγμή που περνάει χάνουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Μέσω τη συνθήκη τη Λισαβόνα, καλώ η κακο ζητηθηκε η εμπιστοσυνη των Ευρωπαίων πολιτών. Με τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ζητήσετε πάλι την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλά η εμπιστοσύνη είναι αμφίδρομη ε, διαδικασία. Δεν μπορείτε μόνο να ζητάτε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και να μην του αποκαλύπτετε την αρχιτεκτονική, τον εσωτερικό μηχανισμό που διέπει τη λήψη των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να ζητούμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών ενώ οι, οι πολιτικοί δεν εμπιστεύονται του πολίτε. Αυτό είναι θέμα δημοκρατία αλλά και σπατάλη γιατί η κοινωνία είναι ένα τεράστιο απόθεμα γνώσεων που θα το κατασπαταλήσουμε αν δεν αναμίξουμε ενεργά τους Ευρωπαίους πολίτες στη διαδικασία ε, λήψης αποφάσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα υπηρετήσουμε την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία υλοποιώντα όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά το γεγονό ότι η διαφάνεια δεν θα είναι μόνο μια ωραία λέξη, αλλά έχει και αυτό περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο του για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική μου τη χώρα και σε άλλες χώρες ε, έχει την φήμη ότι παίρνει τις αποφάσεις ε, μυστικά κατά κύριο λόγο. Γι' αυτό λοιπόν θα υπέθετε κανείς ότι η Κομισιόν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι ανοιχτή και διαφανής. Ανταυτού η Κομισιόν καταθέτει αυτή την πρόταση, τη 1049, ένα κομμάτι της οποίας ε, περιορίζει την πρόσβαση στα έγγραφα που αυτή τη στιγμή είναι δημόσια. Και πέρα από αυτό υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο θυμάμαι τότε που ήμουν στο Χάρβαρτ, που είναι το εξής, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς διαφάνεια και χωρίς ε, τον δημόσιο έλεγχο έχουν μία εγενή τάση να είναι κακές αποφάσεις. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους η Κομισιόν υποβάλει τόσες ε, πολλές ε, αστάθμητες, ε, άστοχες, κακοσχεδιασμένες προτάσεις τις οποίες εμείς στην Αγγλία και άλλες χώρες πρέπει να τις καταπιούμε ένας λόγος είναι η έλλειψη διαφάνειας. Έτσι λοιπόν σε αυτό το θέμα του νομικού πλαισίου καλώ την Κομισιόν να αναθεωρήσει τις σκέψεις της γιατί αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αποφευχθεί μια κακή διαχείριση και κακώς λειτουργούντες οργανισμοί. Πρόεδρε, ο κύριος ε, Γιακολίνο. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την παρέμβαση της Επιτροπής ε, και όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου. Εξάλλου, στο πρόγραμμα της Στεχόλμη επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα πρόσβαση εγγράφων και άλλων οργανισμών ε, της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη της Λισαβόνας ε, επιβεβαιώνει το ίδιο και εγγυάται τον ορισμό των κανονισμών και κριτήρια περιοριστικά για κάθε συγκεκριμένο όργανο ο κανονισμός για τον οποίο ήδη έγινε λόγος ε, έχει εξεταστεί και στο παρελθόν από το Κοινοβούλιο. Ε, σήμερα λοιπόν εκ μέρους όλων υπάρχει συμφωνία ε, για την προσαρμογή του κανονισμού του 2001. Βεβαίως η πρόταση του κυρίου Κάσμαν δεν είναι ικανοποιητική με την έννοια ότι κινείται πέρα από κάθε όριο για έγγραφα τα οποία ε, θα μπορούσαν να είναι καθαρά ε, δημόσιου συμφέροντος. Υπάρχουν και δραστηριότητες ε, για άλλα θέματα. Αυτά όμως όλα πρέπει να διευκρινιστούν ε, για το κατά πόσο πράγματι εκεί πρέπει να επικρατεί διαφάνεια. Γιατί αυτό θα μπορεί να είναι σε αντίθεση με έγγραφα ε, τα οποία προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Εμείς λοιπόν είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε, να ενισχύσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης από πλευράς μεμονωμένων ατόμων. Βεβαίως να επικρατεί ισορροπία όσον αφορά το στόχο. Να διευρυνθεί ο ρόλος ε, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και να υπάρχει μια μεταβατική διάταξη η οποία σιγά σιγά θα μας προσαρμόσει στις ανάγκες του πολίτη έτσι ώστε να υπάρχει συμβασμός με την καλή λειτουργία των οργάνων. Εμείς εμπιστευόμαστε το ρόλο ε, της ΝΙΝ και της μελλοντικής προεδρίας και εμπιστευόμαστε και τις δραστηριότητες επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Δεγιόν, ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ποιο έγγραφο είναι αυτό. Πρέπει να μπορεί κανένας να το βρει ως πολίτης ε, όταν στραφεί προς, τη, ε, προς την ε, Κομισιόν. Αλλά βέβαια κανένας πρέπει να έχει ευγνώητα κείμενα Αυτή είναι η πρωτοβουλία του κύριου Κάσμαν. Και η παρουσίαση είναι πολύ διαφανής ε, εν αντιθέσει με αυτά που είπε η κυρία Ζόμερ. Μπορεί κανένας να έχει ε, πληροφορίες ή άμεσα με ανθρώπινη επαφή ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων για να μπορέσει να πάρει όποια στοιχεία θέλει. Παραδείγματο χάρη, ναι. αν κάποιο ε, ρωτάει πώ λαμβάνονται οι αποφάσει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ λήφθηκαν κάποιε αποφάσει, παραδείγματο χάρη, πριν από την διάσκεψη κορυφή για το κλιματολογικέ αλλαγέ στην Καπερχάγη. Αυτή είναι η πραγματική διαφάνεια. Αυτό θα ήταν καλό. Σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τη δικασία Κάτσο Η κυρία Άπτολα από ό,τι βλέπω ζητάει το λόγο. arvoisa eh, ευχαριστώ πρόεδρε. Το να είναι τα έγγραφα δημόσια σημαίνει ότι ο πολιτή συμμετέχει στι ε, αποφάσεις που λαμβάνονται. Η συνθήκη τη Λισαβόνα θεωρεί ότι αυτό είναι ένα βασικό δικαίωμα των πολιτών. Εάν εμεί δεν προσπίσουμε το δικαίωμα αυτό, ποιος θα το κάνει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα, εδώ, σε αυτή τη συνεδρίασή μα να πούμε ξεκάθαρα ότι είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Δεν επιτρέπεται να υπαναχωρήσουμε, δεν πρέπει να δεχτούμε κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να δεχτούμε αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Υπάρχουν πολλές ε, ε, κακές σε αυτό που συζητάμε εδώ. Δεν θέλουμε εμείς να αντιστρέψουμε κάποιες διεθνεί συμφωνίες, αλλά οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να μάθουν τι συζητιέται με τις τρίτες χώρες που μπορεί ενδεχομένως να άπτε των δικαιωμάτων τους. Δεν θα πρέπει ο καθένας βέβαια να δημοσιεύει όλα του τα, τα γράμματα και τα ταχυδρομεία που έχει. Όταν το θέμα της πρόσβασης ε, των πολιτών στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαφάνεια είναι σημαντική για να μειωθεί ε, η κούραση που έχουν οι πολίτες για τα ευρωπαϊκά θέματα δεν πρέπει να, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Γιατί και εμείς στην ε, Αυστρία βλέπουμε να υπάρχει αυτή η ε, αρνητική στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς επειδή οι πολίτες δεν έχουν την εντύπωση ότι υπάρχει διαφάνεια, ότι δεν έχει καμία πρόσβαση ο πολίτη στην πολιτική. Και τώρα με τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνη και με την εκλογή του Προέδρου του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ΙΠΑ του εκπροσώπου έχει ο πολίτης την εντύπωση ότι δεν έχει καμία δυνατότητα κατανόησης καν και πρόσβεση να παραπάνω για το πώς λαμβάνουν οι αποφάσεις αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε στους πολίτες την ε, ε, εντύπωση ότι μπορούν πραγματικά να κατανοούν τι γίνεται και γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελε κάποιος άλλος, ο Μάικλ Κάρσουμαν, το λόγο. Uh, Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο θέματα. Η κυρία Σόμερ ε, έφυγε βέβαια από την αίθουσα, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω στις σοβαρές κατηγορίες που μου εξακόντησε. Καταρχήν ότι δεν ήμουν διαφανής. Θα ήθελα να πω για τα πρακτικά ότι όλες οι πολιτικές ομάδες και όλοι οι εισηγητές προσεκλήθησαν σε όλες τις συνεδριάσεις. Ακόμη και όταν ήταν απόντες, οι θέσεις τους ακούστηκαν στις συνεδριάσεις αυτές. Όλες ε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν κοινοποιήθηκαν σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές και σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Και μάλιστα έγινε και πρόταση να αποσύρω το ψήφισμά μου γιατί η κυρία Σόμερ το χαρακτήρισε αντιδημοκρατικό και διαφανές και ότι η ομάδα της αγνοούσε τα πάντα για το ψήφισμα αυτό. Πολύ ενδιαφέρον γιατί το απόγευμα είχα διαπραγματεύσει με εκπρόσωπο της ομάδας της για το δικό του σχέδιο ψηφίσματο επί τη προφορική ερώτηση. Άρα φυσικά και το γνώριζε το ΕΛΚ. Ή λοιπόν είναι κακοπληροφορημένη η κυρία Ζόμερ, Οπότε, πραγματικά περιμένω ε, ειλικρινή και καλόπιστη διαπραγμάτευση, όχι μόνο με το ΕΛΚ, αλλά με όλες τις πολιτικές ομάδες. Είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι εδώ, κυρία Βάλστρομ, στην Ολομέλεια. Και σας διαβεβαιώ ότι ούτε εγώ ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε καμία αφιβολία για την προσήλωσή σας προς το άνοιγμα και τη διαφάνεια. Είχατε δίκιο ότι ο καθένα έδωσε τη μάχη για το θεσμικό του όργανο. Και εσεί πραγματικά δώσατε τη μάχη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με υποδειγματικό τρόπο και ουδέποτε δεν, δεν προδώσατε τι αρχέ ε, τη διαφάνεια και του ανοίγματο. Είστε και θα παραμείνετε ε, μια καταπληκτική υπάλληλος ε, της δημόσιας ε, υπηρεσίας, λειτουργός, ε, αξιοπρεπής, δίκαιη, έντιμη, ειλικρινής και ως, και ένας από τους ανθρώπους που είχαν το προνόμιο να έρθουν σε επαφή μαζί και να σας γνωρίσουν από κοντά θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα άλλος κανεί το λόγο στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye. Όχι, οπότε να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Μάρστρο, στην Υπουργό Μάλστρομ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κοινοτική νομοθεσία για την πρόσβαση στα έγγραφα και η οδηγία 1049 είναι μια οδηγία που γνωρίζουμε καλά και με τον Μάικλ Κάσμαν και την ε, κυρία Βάλστρομ συμβάλαμε στην ε, διαμόρφωση αυτής της οδηγίας. Η συνθήκη της Λισαβόνας μάλιστα μας επιτρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι και να πάμε ακόμη πιο μακριά. Γιατί η εμβέλεια αυτού του κανονισμού 1049 ενισχύεται και διευρύνεται. Χρειάζεται διοργανικό διάλογος και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιμέναμε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι και η Ισπανική Προεδρία θα περιμένει το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσει να συνεχίσει τις διοργανικές επαφές. Πάντως και στο ενδιάμεσο διάστημα δεν μείναμε τα χέρια σταυρωμένα. Είχαμε πολλές συναντήσεις, μία σήμερα το πρωί, όπου καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα έγγραφα και θα πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα να διευκολύνουν την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στα έγγραφα. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε και τον ιστοτοπό μας, ώστε οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες να παρακολουθούν την ομοπαρασκευαστική διαδικασία ενός κειμένου από τη στιγμή της πρότασης ε, από την, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τη στιγμή της έγκρισης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Έτσι θα βελτιωθεί η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα πράγματα είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά και θα μας επιτρέψουν να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και να μειώσουμε τις υπόνοιες περί αδιαφάνειας. Γιατί αν δεν βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών θα πλήξουμε την ομιμότητα των αποφάσεών μας. Ελπίζω ότι ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί όχι βέβαια κατά τη διάρκεια τη Σουηδική Προεδρία που τελειώνει, αλλά στι επόμενε Προεδρίε και ευχαριστώ θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον εισηγητή, τον κύριο Κάσμαν. Η κυρία Επίτροπο ε, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, αυτός πράγματι ήταν ε, ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο ε, να με συγκινήσετε και πού θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο θέμα για να έχω μάλλον την τελευταία μου παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλύτερο θέμα από το, τη διαφάνεια και το άνοιγμα δεν υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μία πρόταση. Είναι η μόνη πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό το πράξαμε στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναπομπής. Άρα δηλαδή οι αρχές που διέπουν αυτόν τον οργανισμό είναι ε, σωστοί. Βεβαίω ε, πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις διατάξεις, να είναι περισσότερο αποτελεσματικέ. Αυτή είναι η ιδέα που υπήρχε πίσω από την αναπομπή. Έχουμε διαφορετικές απόψεις ε, για το πώς πρέπει να ορίζονται κάποια έγγραφα, όμως ε, αυτές εξακολουθούν να είναι διαπραγματεύσεις στις οποίες πρέπει να συμμετέχουμε για να διασφαλίσουμε την πρόοδο. Και για να τα κάνουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε την πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα από δικής μας πλευράς και επίσης πιστεύουμε ότι με βάση τη νέα συνθήκη μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας ε, επεκτείνοντας ε, το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Και κατά την άποψή μας ε, από πλευράς Επιτροπής αυτή είναι η βασική διαφορά. Τώρα πλέον θα καλύπτονται όλοι οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα. Ξεκολουθούμε να ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα προσφέρει το συντομότερο δυνατόν μια πρώτη ανάγνωση. Θα έχουμε και την άποψη του Συμβουλίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις απαραίτητες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε κάποια στιγμή σε απόφαση. Υπάρχει μια σειρά σημαντικών θεμάτων που θίξατε κύριε Κάσμαν και εσεί ε, στην έκθεσή σας και υπάρχουν ε, και άλλοι τρόποι να χρησιμοποιήσουμε αυτά που λέτε γιατί είναι λιγάκι εκτός πεδίου εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Όμως εξακολουθούν να είναι σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με τα Μητρώα και με όλα αυτά ε, που συζητήσαμε σήμερα. Πράγματι μπορούμε να βελτίσουμε το άνοιγμα, τη διαφάνεια και με άλλες ε, μεθόδους, όχι μόνο μέσα από τον κανονισμό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, ξέρετε ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά εγώ παρόλα αυτά ανέλαβα την πρωτοβουλία να καταρτήσω ένα πρόγραμμα δράσης για το άνοιγμα που συζητήθηκε σήμερα. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συνεχίσουμε για το άνοιγμα και τη διαφάνεια, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Και με αυτή την ε, χαρούμενη κατακλίδα, γιατί εγώ ήθελα ε, να επικρατεί έτσι ένα ευχάριστο περιβάλλον. Να σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και να σας ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Επιτρέψτε μου και εγώ να δράξω την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το πνεύμα συνεργασία που επιδείξατε όλα αυτά τα χρόνια και σε εσά καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Κλείνει λοιπόν συνάδελφοι η συζήτηση για αυτό το θέμα. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Πέμπτη. Επόμενο θέμα στην ε, ημερήσια διάταξη είναι οι δηλώσεις ε, της ε, Κομισιόν και του Συμβουλίου για την κατάσταση στη Γεωργία.